Δίνω το λόγο στην κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φτάνουμε στην ε, τελική φάση μιας εργασίας η οποία έχει χρειαστεί πολλούς μήνες για να καρποφορήσει. Η επιχειρηματία των γυναικών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και φυσικά είναι κουραστικό να το ακούει κανείς, αλλά είναι κάτι που επλήγει ιδιαίτερα από την χρηματοπιστωτική ε, κρίση. Θέλω να ευχαριστήσω του κοιόδης για τη βοήθειά τους σε όλες τι φάσει αυτή της έκθεση. Έχουμε φτάσει σε μια στρατηγική η οποία <clears throat> έχει σαν στόχο να συναθρήσει όλες τι πολιτικές ομάδες γύρω από μια κοινή θέση, μια θέση εγκάρσια η οποία περιστρέφεται γύρω από μια κοινή προσέγγιση. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέρφους για την κοινή θέλησή τους να γίνουν οι γυναίκες πρωταγωνίστρες της οικονομικής ανάκαψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μελετήσει, έχουμε αναλύσει, ανατάμει τους λόγους που αποτελούν τους εξωτερικούς παράγοντες που οδηγούν σε προσκόμματα στο επιχειρήν των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει μονάχα 30% επιχειρηματίες γυναίκες. Η διαδικασία κυραφέτησης των γυναικών στους προηγούμενους αιώνες που οδήγησε σε πολύ σκληρές ε, μάχες και αγώνες για να εξασφαλιστεί η ισότητα των δύο φύλων δεν έχει φτάσει ακόμα στο τελικό τη στάδιο, δεν έχει επιτύχει την ισότητα στον τομέα του επιχειρής. <clears throat> Μεταξύ των εμποδίων που έχουμε αντιμετωπίσει είναι αυτό που και αυτό που μας οδήγησε στην έκθεση αυτή είναι λόγοι οικονομικοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί. Οι γυναίκες πολλές φορές είναι θύματα πεπαλαιωμένων στερεοτύπων, θεωρούνται ότι μόνο δευτερό δεύτερου επίπεδου ρόλους μπορούν να διαδραματίσουν. Οι γυναίκες πρέπει να σκέφτονται την οικογένεια, τα παιδιά, τους γέρους, την οικογένεια, λες και η μητρότητα είναι ένα εμπόδιο και όχι η κορύφωση της αξιοπρέπειάς τους. Οι οδηγίες μας λένε ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση βάση του φύλου, αλλά στην πραγματικότητα η πρόσβαση στην ε, ισότητα σε ό,τι αφορά την παροχή των υπηρεσιών δεν υπάρχει. Οι γυναίκες είναι θύματα διακρίσεων όταν θέλουν να πάρουν χρηματοδότηση. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους νέους μας στο πνεύμα του επιχειρήν, της ανάληψης κινδύνου, της ανεξαρτησίας και της δημιουργία επιχειρήσεων. Το κείμενο που θα ψηφίσουμε αύριο εστιάζει σε πέντε βασικούς θεματικούς τομείς. Πρώτα απ' όλα, το κύριο θέμα είναι η ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής ζωής και επαγγελματική ζωή, που δυστυχώς είναι ένα από τα κύρια εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στην Ευρώπη όταν θέλουν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. <clears throat> Προτείνουμε εδώ να υπάρξει μια πραγματική ορθολογικοποίηση της δυνατότητα του να είναι διαθέσιμα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, υποστήριξη για ε, φροντίδα των ηλικιωμένων και babysitting για τα παιδιά. Δεύτερον, μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών από δίκτυα εκπαίδευση στον επιχειρηματικό τομέα. Όλα αυτά είναι σημαντικέ ψηφίδε για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για, το επιχειρήν των γυναικών. Το πραγματικό <clears throat> εμπόδιο το τρίτο μεγάλο εμπόδιο είναι η πρόσβαση στα, στη χρηματοδότηση των γυναικών. Εδώ χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην πρόσβαση υπηρεσιών. Οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίζουν όλους με τον ίδιο τρόπο και όχι να δίνουν προτίμηση στα ανδρικά σχέδια επενδύσεων. Επίσης πρέπει να υπάρξει μια κουλτούρα του επιχειρήν στα να ενσταλλαχθεί στα παιδιά μας και να δώσουμε λοιπόν στα κορίτσια και τις κοπέλες τη δυνατότητα να μπουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση. Και τέλος, οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εργάζονται όχι μόνο στου κοινωνικού τομείς, αλλά και στου τομεί που ενάπτονται με τις νέες τεχνολογίες και την πράσινη οικονομία. Έχουν κλείσει λοιπόν τα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου. Θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους συναδέλφους αύριο να υπερψηφίσουν αυτό το ψήφισμα υπέρ μιας Ευρώπης η οποία θα είναι <clears throat> πιο ενσωματωμένη. Τελειώνω με τα λόγια της Οριάννα Φαλάτσι. Το να είναι κανείς μια γυναίκα είναι κάτι το οποίο είναι εγωιτευτικό, είναι μια περιπέτεια που θέλει θάρρος, μια πρόκληση που δεν τελειώνει ποτέ. Ζητώ από τους συναδέλφους λοιπόν να ε, αγωνιστούν μαζί μου για αυτή την περιπέτεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ματέρα. κυρία Γκάλπε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια στην κυρία Ματέρα. Εξαιρετική έκθεσή της. Ευχαριστούμε. Πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες ε, ε, να ακολουθούν επιχειρηματική καριέρα περισσότερο. Αυτό θα βοηθήσει και την οικονομική ανάπτυξη αλλά θα είναι πολύ σημαντικό και για τις ίδιες τις ε, γυναίκες ε, για να ευοδοθούν ε, οι ανησυχίε τους στα όνειρά τους. Θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε, να φτιάξουν, να οικοδομήσουν τις επιχειρηματικές τους καριέρες, την επιχειρηματική τους σταδιοδρομία. Ασφαλώς υπάρχουν εμπόδια, τα ανέφερε η κυρία Ματέρα. Ένα πολύ σημαντικό είναι η πρόσβαση χρηματοδότηση. Θα πρέπει οι συνθήκες να ευνοούν την πρόσβαση αυτή. Επίσης θα ήθελα να στηρίξω την ιδέα του, της δικτύωσης. Είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικές για την οικονομία ασφαλώς, αλλά δεν είναι το μοναδικό εργαλείο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Δεν είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε για να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Πιστεύω ότι η έκθεση πάντω είναι πολύ καλή, πολύ θετική, την στηρίζω και θα την υπερψηφίσω αύριο. Κύριε Πρόεδρε, η προσέγγιση για την ισότητα των ε, φύλων προϋποθέτει και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στα κράτη-μέλη τα προώθηση δηλαδή πολλαπλών δράσεων για την υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Ε, θα πρέπει να πλουστευτεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και άλλες μορφές ε, υποστήριξης, μείωση της γραφειοκρατίας, απάλληψη άλλων εμποδίων ε, στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Τα κράτη-μέλη αναθεωρούν ε, ε, τα μέτρα τους ε, για να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που ενημερώνουν ε, τις επιχειρηματίες εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και φροντίζουν για επιτυχή στα διοδρομία. Θέλω να συγχαρώ τέλος την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Κυρία Τόμασικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το επιχειρήν και η προσέγγιση, η σωστή προσέγγιση προς τις επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρυνθούν στην παιδεία και την κατάρτιση σε όλες τις ηλικίε και στα δύο φύλλα. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί και να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση. Το επιχειρήν είναι πολύ λιγότερο διαδεδομένο μεταξύ γυναικών και από ό,τι μεταξύ ανδρών. Έχει μεγάλο δυναμικό να αναπτύχθει περισσότερο, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω τις προτάσεις που ζητούν από τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθορίσουν πολιτικές για ισορροπία ιδιωτικής και επαγγελματική ζωής. Αυτό δεν είναι η δουλειά των πολιτικών και των θεσμών. Η κάθε οικογένεια έχει τη δική της αυτονομία. Σε κάθε οικογένεια πρέπει η γυναίκα και ο άντρας να πάρουν τις αποφάσεις τους για το καλύτερο συμφέρον των παιδιών. Οι πολιτικοί λοιπόν δεν πρέπει να μπουν στα χωράφια αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπιλμπάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ματέρα για την ε, δουλειά σας η επιχειρηματικότητα, η αυτοπασχόληση ε, των γυναικών είναι μια πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας η οποία χαρακτηρίζεται από ανισότητα. Οι γυναίκες θεωρούν ότι η αυτοπασχόληση και η επιχειρηματικότητα είναι λιγότερο ελκυστικές από ότι οι άντρες. Ε, αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη χρηματοδότηση και ε, εργάζονται σε εργασίες που έχουν μικρότερη προσθέμενη αξία η γυναικεία συνεισφορά ε, δεν εκμεταλλεύεται όλων των δυνατοτήτων και η κοινωνία χάνει ταλέντα και ευκαιρίες. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε αντικειμενικά δεδομένα τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε καλύτερη διάγνωση, συγκεκριμένες πολιτικές, τη χρηματοδότηση, ε, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εκπαίδευση. Ε, επίσης να συνεχίσουμε να πολεμάμε τα στερεότυπα η, η ανισότητα δεν βλάπτει μόνο τις γυναίκες. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα, αν το πιστεύουμε. Η ανισότητα, κύριε Επίτροπε, μας, κάνει να χάνουμε, μας βγάζει χαμένους όλους. Ευχαριστώ. Κύριος Βέγγας, μετά από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές είναι φανερό ότι η, ε, η ένδια, η ανεργία και όλα αυτά έχουν γυναικείο πρόσωπο και ο αποκλεισμό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Με το να το αντιμετωπίσουμε αυτό θεωρώντας το επιχειρήν σπανάκια πανάκια είναι λαθασμένο. Θα πρέπει να μην προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια με κάτι που την κάνει χειρότερο. Πρέπει να έχουμε μια νομοθεσία η οποία θα εξασφαλίσει την ε, απασχόληση ποιότητος και με αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να προωθούμε την επισφαλή εργασία που κυρίως ασκείται από τις γυναίκες. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες όλες οι γυναίκες να είναι πλήρεις πολίτες, ισότιμοι. Αυτό σημαίνει ασφάλεια στον χώρο εργασίας, χωρίς διάκριση μεταξύ των φύλων και δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας που μπορούν να εξασφαλίσουν την υγειονομική περίθαλψη και την παιδεία για όλα τα παιδιά. Δυστυχώ δεν είναι αυτή η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον αγώνα των γυναικών και των εργαζομένων, όμω κάπου θα το καταφέρουμε. Quiero comentarles que hemos tenido. Eh, eh, είχαμε διπλάσια αιτήματα από θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε σε πέντε λεπτά. Προσπαθήσαμε πάντως και νομίζω το καταφέραμε να μιλήσει ένας εκπρόσωπος από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε άλλους ετούντες. Όλες οι ομάδες πάντως πήραν το λόγο. Ο λόγος στον κύριο Επίτροπο. Mr. President, thank Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ματέρα. Όπως ακούσαμε και όπως γνωρίζουμε, οι μικρομεσαίες Επιχειρήσει θα είναι η ατμομηχανή για την δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη και θα ξεκλειδώσουν το πλήρε δυναμικό τη οικονομία μα. Γι' αυτό όμω χρειάζεται να ξεκλειδώσουμε την δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό όλου του πληθυσμού, άντρων και γυναικών. Γνωρίζουμε ότι η επιχειρηματικότητα όμω ε, ελκύει λιγότερο τι γυναίκε από του άντρε, 63% των γυναικών λένε ότι δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό του να ξεκινήσουν δική του επιχείρηση. Ε, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 52% στου άντρε και όπως ακούσαμε ένα από τα βασικά εμπόδια ε, είναι τα στερεότυπα, ε, έλλειψη αυτοπεποίθησης και δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε επιχειρηματικά δίκτυα. Γι' αυτό το λόγο ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός και έχει νόημα τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν και την επιχειρηματικότητα ε, ως μάθημα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Οι γυναίκες είναι, διαφέρουν όχι μόνο ως προς, ε, την, ως προς αυτό που τις εμπνέει, αλλά και ε, είναι διαφορετικές και στον τρόπο που διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους. Για παράδειγμα, μετρούν καλύτερα και ε, πιο προσεκτικά τους κινδύνους. Γι' αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις των γυναικών είναι πιο βιώσιμες γενικά από αυτές των ανδρών. Στην αρχή όμως ε, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, για να εξασφαλίσουν τα κεφάλαια κίνησης. Πώς θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε με ειδικά ενδεχομένως προγράμματα ε, για τους επενδυτές έτσι ώστε να καταλάβουν τον επιχειρηματικό ρόλο των γυναικών. θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στις γυναίκες υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες ε, έτσι ώστε να τις διευκολύνουν και μέσω των ε, δικτύων γυναικείας επιχειρηματικότητας και συμβούλων, ε, μεντόρων. Ε, εμείς θα ξεκινήσουμε μια πλατφόρμα για γυναίκες όλων των ηλικιών που θέλουν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Αυτή η πλατφόρμα θα δίνει συμβουλές, εκπαίδευση και δυνατότητες δικτύωσης για τις γυναίκες. Θα είναι ε, μια μονοπευθυντική θηρίδα για τις γυναίκες επιχειρηματίες. Θα τους επιτρέπει να έρθουν σε επαφή με άλλες οργανώσεις, με άλλα δίκτυα και να αναζητήσουν πληροφορίες για χρηματοδότηση. Χάρη σε ένα πυρωτικό project του Χρηματοδοτητού Κοινοβούλιο θέλουμε να εξασφαλίσουμε και εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω επιχειρηματικών αγγέλων γυναικών. Ε, επίσης σημαντικός ο ρόλος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μέσω της ομάδας ε, εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα η Κομισιόν εργάζεται έτσι ώστε να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών στι κοινωνικέ επιχειρήσει στην Ευρώπη. Τέλο, η υποστήριξη τη γυναικείας επιχειρηματικότητα σημαίνει και τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντο μέσα στο οποίο να εκμεταλλευτούν τι ικανότητέ του στο μέγιστο. Γι' αυτό το λόγο θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να διευκολυνθεί ε, ε, η, φροντίδα των ηλικιωμένων και των παιδιών, έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι γυναίκες. Η Ευρώπη χρειάζεται τα ταλέντα όλων των πολιτών της και η Κομισιόν σας βεβαιώνω ότι θα συνεχίσει έτσι ώστε να υποστηρίζει τη γυναική επιχειρηματικότητα. Και η έκθεση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μας βοηθήσει σε αυτό μας το καθήκον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Πλούρα για τις ε, πολιτικές